αγαπητή Επίτροπε, αγαπητή Σεσίλια. Άρχεται η σημερινή συνεδρίαση με πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη μια προφορική ερώτηση για τις διακρίσεις λόγω κάστας. Επιτροπή Ανάπτυξης είναι η επιτροπή που έχει καταθέσει αυτή την προφορική ερώτηση. Από ό,τι βλέπω όπως είναι λογικό άλλωστε, είναι η Εύα ε, Ζολή, η οποία έχει ως ε, συντάκτρια προφορικής ερώτησης πέντε λεπτά. Εύα, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε και είπατε πρόσωπε, αγαπητοί συνάλφοι, Απαρτχάιντ είναι ο όρος που πέραν του καθεστώτος ε, αντικατοπτρίζει και ταπεινώσεις βία χρησιμοποιήθηκε το 2006 από τον τότε Ινδό Πρωθυπουργό Σιγκ για να μιλήσει για την κατάσταση των άθικτων ε, στη χώρα του. Παρά όμως αυτή την πολύ ε, σοκαριστική δήλωση και την κατάργηση αυτής της ε, ιδιότητας του άθικτου και παρά τους διάφορους νόμους 200 ε, εκατομμύρια άνθρωποι, άνδρες και γυναίκες ε, σπασμένοι, ντάλιτ, ε, υποφέρουν σε καθεστώς πλήρους ατιμορρησίας. Από το 2005 από το 2001 2005 στην Ινδία, τρεις γυναίκες ντάλιτ κάθε, βιάζονταν κάθε ημέρα. Κάθε 18 λεπτά είχαμε μια αξιόπινη πράξη κατά ενός ντάλιτ. Το Πακιστάν έχει υπογράψει την Κομμουνική Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ωστόσο εκατομμύρια πολιτών του δεν χαίρουν των δικαιωμάτων των ελευθεριών που διακηρύσει αυτή η ε, διακήρυξη, ακριβώς ε, λόγω της γέννησής τους. Θα ήθελα λοιπόν ε, να δούμε αυτές τις διακρίσεις λόγω κάστας για μια ακόμη φορά και για την απάνθρωπες και γιατί αντιβαίνουν στο διεθνέ Δίκαιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και γιατί είναι και ένα μίσον δομικό παράγοντα για τη φτώχεια και τι ανισότητε που επικρατούν. Το apartheid αυτό έχει οικονομικέ, ε, φρικτέ κοινωνικο οικονομικέ επιπτώσεις αρνούνται στους ανθρώπους αυτούς ανώτερα κλιμάκια και θέσεις εργασίας. Τους αρνούνται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι αστυνομικές υπηρεσίες όταν δεν τα παραβιάζουν. Μόνο 10% των γυναικών τάλιτ εκπαιδεύονται, μορφώνονται. Η έξοδος από την ε, ε, φτώχεια καταλαβαίνουμε ότι για πολλές είναι κάτι αδύνατον. Είναι μεν η Ινδία αναδυόμενη χώρα, αλλά αυτό το φαινόμενο δεν φαίνεται να εκριζώνεται το αντίθετο. Το χάσμα μεταξύ των Τάλιτ και μη Τάλιτ από τις αρχές της δεκαετίας του 90 διωγγώνεται. Και έτσι αποδεικνύεται η αποτυχία της αναπτυξιακής πολιτικής που αγνοεί πολύ συχνά αυτό το πρόβλημα. Καμία βούληση δεν υπάρχει φαίνεται από τους ηθήνοντες στη χώρα που ναι μεν έχουν ε, κάποιες, κάποια από αυτούς προωθήσει κάποιους νόμους για θετική διάκριση που δεν πέτυχαν όμως. Και θα πρέπει και εμείς στην Ευρώπη να αναγνωρίσουμε αυτές τις διακρίσεις λόγω κάστας ως μια διακριτή μορφή διακρίσεων που είναι πολύ έντονη και στο κοινωνικό και στο θρησκευτικό επίπεδο. Τα θύματα αυτού του διαχωρισμού λόγω κάστας ε, θα μπορούσαν έτσι να λαμβάνονται υπόψη καλύτερα και στα αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αποτελεσματικότητα της ε, βοήθειας ε, έτσι θα ενισχυθεί. Η συνοχή, η συνεκτικότητα των εξωτερικών πολιτικών με την αναπτυξιακή πολιτική επιβάλλει όχι μόνο την αξιολόγηση σε περίπτωση που έχει αυτή η κατάσταση, εμπορικέ ε, και άλλε συμφωνίε Ευρωπαϊκή Ένωση με τι χώρε αυτέ, αλλά απαιτείται πέραν αυτού και η ενσωμάτωση ρήτρα ε, για τις διακρίσεις ε, λόγω Τα πρόσφατα γεγονότα στο Παγκλαντέ. σε εμά του Ευρωπαίου δεν μα επιτρέπουν πλέον να δηλώνουμε άγνοια. Οι ευρωπαϊκέ επιχειρήσει άμεσα ή έμεσα συμμετέχουν σε αυτή την κατάσταση που οδηγούν ορισμένους ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν ενδεχομένως στη, στο κοινωνικό επίπεδο, στο κοινωνικό στρώμα που έπρεπε να ε, αντιμετωπίζονται ως σκλάβοι. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε όλες ε, τις δυνατότητες που μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθήσουμε κοινές πρωτοβουλίες με στόχο την ε, εκρίζωση των διακρίσεων λόγω μια ε, διάκριση ε, είναι πάντα διάκριση και πρέπει να ξέρουμε ότι έχουμε και εμείς ευθύνες να προστατεύσουμε και να προβάλλουμε τα δικαιώματα των ανθρώπων που, είναι, που υφίσταται τη διακριτική μεταχείριση ε, και είναι απομονωμένοι, εξωστρακισμένοι στο ευρωπαϊκό επίπεδο. οι διακρίσεις αγνοούν τα σύνορα η Ρωμά είναι ένα πολύ ευλωτό παράδειγμα που σε πολλά κράτη-μέλη υφίστανται το ρατσισμό, τις προκαταλήψεις, τις διακρίσεις. Είναι εκτός του οικονομικού πολιτικού βίου, εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος και του συστήματος υγείας. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις τρίτες χώρες να ξεκινήσει ειλικρινείς επικοδομητικές συνομιλίες για να τεθεί τέρμα σε κάθε μορφής διάκριση που αποτελεί τροχοπέδι για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ κυρία Ζολή, κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Επίτροπο, στην κυρία Μάλστρομ, για να απαντήσει στην προφορική ερώτηση της κυρίας Ζολή, εξ ονόματος Επιτροπής Ανάπτυξης. Αγαπητή Σεσίλια έχεις το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Ζολή που υπέβαλε αυτή την υπόθεση έτσι ώστε να μπορέσω κι εγώ εκ μέρους της ΕΠΑ της εκπροσώπου να μιλήσω για το θέμα αυτό της διάκρισης σε διάφορες κοινωνίες. Έχουμε δεσμευτεί να αντιμετωπίσουμε κάθε είδους διακρίσεις ο αγώνας αυτός είναι μια προτεραιότητα ανθρωπίνων δικαιωμάτων για το ευρωπαϊκό στρατηγικό πλαίσιο και το σχέδιο δράσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ε, διακρίση με βάση την κάστα είναι κομμάτι αυτού. Τα κράτη-μέλη έχουν χρησιμοποιήσει πάρα πολλά μέτρα όπως ε, διμερής διάλογος, ε, οικονομική ενίσχυση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η παρέμβαση διαφόρων οργανισμών. Επίσης ε, αυτό το θέμα ε, περιλαμβάνεται συνεχώς στους διαλόγους μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα και στι επαφέ μας με όσους ε, αυτών. Επίσης ε, και με τις χώρε εταίρου συζητούμε τα θέματα αυτά όπως η Ινδία, το, το Νεπάλ, το Μπαγκλαντέ, το Πακιστάν αλλά και η Μαυριτανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη έτσι ώστε να καταργηθεί η διάκριση με βάση την κάστα και οι επιρροές της μέσω των ευρωπαϊκών εργαλείων, όπως αυτό για τα, ευρωπαϊκά, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Το εργαλείο αυτό και τα σχετικά στρατηγικά έγγραφα από το 2011 το 2013 περιλαμβάνουν σαφείς αναφορές σε διακρίσεις με βάση την κάστα. Για παράδειγμα, στην Ινδία οι διακρίσεις με βάση την κάστα θεωρούνται ε, οριζόντιο ε, θέμα που, έχει πάρα πολλές, ε, που προκαλεί πάρα πολλέ ανησυχίε και έχουν υπάρξει πάρα πολλές προτάσεις ως προ αυτό. 4 εκατομμύρια χρηματοδότηση δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της βίας κατά των κοριτσιών και των γυναικών. Επίσης, Έχουμε μια πολύ προσέγγιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επίσης και για τι οικονομικες οικονομικε και ψυχολογικές, ψυχολογική βοήθεια προ τα θύματα έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους ε, παράχουμε πρόσβαση στην, στην ε, εκπαίδευση, στα εργασιακά δικαιώματα. Στον Μπαγκλαντές η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, χρηματοδοτεί πάρα πολλά project για τη μείωση της φτώχειας και προστασία των πιο φτωχών και εξαφλαιωμένων ομάδων. Επίσης, χρηματοδοτούμε project που έχουν να κάνουν με πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα θύματα της διάκρισης με βάση τη βία. Και αυτό έχει να κάνει και σε αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει 30 εκατομμύρια ευρώ στο Μπαγκλαντές και στο Πακιστάν ε, για την βελτίωση της πρόσβασης και της λειτουργίας των τοπικών δικαστικών και αστυνομικών συστημάτων. Σε σχέση με την ανθρωπιστική βοήθεια να πω ότι πάντα ε, δεν είναι βασισμένη σε διακρίσεις. Προφανώς βασίζεται στις ανάγκες και δίνεται ιδιαίτερη σημασία στις πιο ευάλωτες ομάδες. Οι ανθρωπιστικέ δράσει που, που χρηματοδοτούνται συγγνώμη, από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στην Νοτιοανατολική Ασία βασίζονται ακριβώ σε προγράμματα που έχουν, που έχουν ω στόχο την αντιμετώπιση τη διάκριση με βάση την κάστα σε, πολύ, σε επίπεδο έχουμε συμβάλει ε, στη δουλειά που έχει γίνει από την υποεπιτροπή του ΟΗΕ για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης συμβάλλουμε στη συζήτηση που έγινε για τις διακρίσεις με βάση την κάστα στην, ε, διαδικασία περιοδικής αναθεώρησης ε, του ΟΗΕ για την ιδέα των Πακιστάν, τη Σιρλάνκα, τον Μπαγκλαντές. Τέλος, οι διακρίσει με βάση την κάστα αποτελούν προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε να τι αντιμετωπίσουμε και το κάνουμε με τον πιο συνακτικό και αποτελεσματικό τρόπο ω τμήμα τη γενική μα στρατηγική κατά οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδου διάκριση. Έχουμε εργαλεία, έχουμε μέσα στα χέρια μα. Έχουμε διμερείς διαλόγους, για παράδειγμα, οικονομική ενίσχυση ε, των οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών. Χρησιμοποιούμε την ευελιξία και με μια προσέγγιση που ταιριάζει στη χώρα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Σε ευχαριστώ, Σεσίλια. Γνωρίζουμε τη δέσμευσή σου και είμαστε βέβαιοι ότι θα κάνεις πάντο δυνατόν για το τόσο σημαντικό, τραγικό αυτό ζήτημα. Περνάμε στο γύρο των ομιλητών, με πολιτικέ ομάδε. Κατά πρώτον, το λόγο έχει για δύο λεπτά εκ μέρους του ΕΛΚ ο συνάδελφος Σβένσον. Ε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στα δικτατορικά καθεστώτα υπάρχει σαφώς καταπίεση των ε, πολιτών. Αυτό το γνωρίζουμε σε χώρες όπου θα ελπίζαμε όμως να υπάρχουν δημοκρατικοί θεσμοί και δομές καθώς και να γίνονται σεβαστές οι δημοκρατικές αξίες, τέτοια φαινόμενα είναι απαράδεκτα. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει να συζητηθεί και πρέπει να συζητάτε ε, όποτε προκύπτουν τέτοια ζητήματα. Είναι ένα θέμα που συχνά το έχουμε επαναφέρει στην ημερήσια διάταξή μας, ε, τη διακριτική μεταχείριση λόγω κάστας. Υπάρχουν χώρε που φέρονται με διαφορετικό τρόπο σε ένα μέρο του πληθυσμού του γιατί του έχουν ορίσει ω ανέγκυχτου. Μιλάμε για το μισό πληθυσμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση αν συγκρίνουμε τι τάξει μεγεθών. Δεν μπορούμε λοιπόν να μιλάμε για παραδόσει ηθικά έθιμα για να εξηγήσουμε τέτοιου είδου συμπεριφορέ. Οι νοοτροπίε πρέπει να αλλάξουν. Εάν θέλουμε να έχουμε εμπορικέ σχέσει ή άλλου είδου σχέσει θα πρέπει να δοθεί έμφαση από το πρόβλημα. Το βρίσκω απαράδεκτο να βλέπουμε γυναίκες και παιδιά ουσιαστικά να κλείνονται σε κλουβιά από τα οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν. Πρόεδρε, χαίρομαι ιδιαίτερα που τέθηκε αυτό το ερώτημα και που περιλήφθη στην ημερήσια διάταξη, αλλά Ας μην σταματήσουμε στη συζήτηση τη σημερινή, μια πέμπτη πρωί στο Ευρωκοινοβούλιο απλώς, να πιέσουμε για να δοθεί σημασία στα ε, θέματα αυτά. Τα συγκεκριμένα κράτη έχουν προσυπογράψει στη χάρτα του ΟΗΕ για την ανεξιθρησκεία, την ελευθερία της έκφρασης, την ελευθερία των ε, θρησκευτικών πεπιθήσεων όμως έτσι ε, απογοητεύουν τους πληθυσμούς τους. Θα πρέπει λοιπόν αυτού του είδους διακριτική μεταχείριση να ε, γίνει αντικείμενο καταγγελίας ως κάτι απαράδεκτο. Πρόεδρε, πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα, ώστε να μπορέσουν οι δημοκρατικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες να προστατευτούν και αλλού. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε, κύριε Σβένσον. Εκ μέρου ε, των συναδέλφων των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριο Μάικλ Κάσμαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που προεδρεύετε εσεί όταν μιλάμε για θεμελιώδεις αξίες. Θα ε, συμφωνήσω απολύτω με την εισαγωγική παρέμβαση τη κυρία Ζολή και της, του κυρίου Σβένσον. Δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, καμία θέση ε, για διακριτική μεταχείριση λόγω κάστα στι εξωτερικέ και εσωτερικέ σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση και ελπίζω σήμερα να αποστείλουμε ένα ισχυρό μήνυμα. Κυρία Επίτροπε, γνωρίζω τι δεσμεύσει σα, ξέρω την αίσθηση ευθύνη που έχετε και ακούω τι είπατε, αλλά πρέπει να πω ότι δεν έχουμε πετύχει τίποτα. Εάν έχουμε κάνει όλε αυτέ τι προσπάθειε, έχουμε όλα αυτά τα εργαλεία και 220 εκατομμύρια άνθρωποι ακόμη είναι θύματα διακριτική μεταχείριση μόνο και μόνο λόγω τη ε, προέλευσή του από μια συγκεκριμένη κάστα και του γεγονότο ότι ανήκουν σε μια συγκεκριμένη κάστα, Όλες οι συμφωνίες μας, εμπορικές, σύνδεσεις, δεν μπορούν να προχωρούν. Θα πρέπει να υπήρχε μια διαπραγμάτευτη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όλες μας οι σχέσεις ε, να ε, εξετάζουν και αυτό το ζήτημα. Το αν υπάρχει διακριτική μεταχείριση ε, λόγω κάστας. Όταν αγοράζουμε από το Πακιστάν, την Ινδία, τον Μπακλαντές. Όταν ουσιαστικά κάνουμε φτωχότερους τους ανθρώπους αυτούς, στις πλάτες τους κερδίζουμε, στις ε, και ακριβώς πίσω από την πλάτη τους ε, συμμετέχουμε στην διακριτική μεταχείριση εναντίον τους. Μιλάμε για μια συνθήκη προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που έχουμε προσυπογράψει. Μιλάμε για κορίτσια, γυναίκες που είναι θύματα βίας, ε, κακομεταχείρισης. Μόνο και μόνο με το πρόσχημα ότι ανήκουν σε μια διαφορετική κάστα. Προ το τέλο τη θητεία μα, λοιπόν, χαίρομαι ιδιαίτερα που ενώθηκαν εδώ όλε οι πολιτικέ ομάδε για να πούν ότι όχι, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αλλά να πω και δημοσίω και να πω και στου πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε από πού αγοράζουμε τα προϊόντα μα. Διότι όταν αγοράζουμε πουκάμισα, γραβάτε και παπούτσια από τέτοιε χώρε, Εάν στι χώρε αυτέ δεν γίνονται σεβαστά τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και ασκείται διακριτική μεταχείριση με σκανδαλώδη τέτοια προσχήματα όπω αυτό τη Κάστας, τότε θα πρέπει ε, μεμονωμένα να τι απομονώνουμε και να μην έχουμε εμπορικέ σχέσει μαζί του. Σε ευχαριστώ, Μάικλ. Εκ μέρου των ε, Φιλελεύθερων Δημοκρατών, για δύο λεπτά έχει το λόγο ο κύριο Ντόνσκι. Πόνε Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Οι διακρίσει λόγω κάστα είναι ένα από τα μεγαλύτερα παράδοξα του 21ου αιώνα. Έχει γίνει μικρότερο ο κόσμο μα, ο πλανήτη μα. Έχουν σχεδόν καταργηθεί τα σύνορα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά εκατομμύρια ανθρώπων οι οποίοι δεν χαίρουν κανένα σχεδόν δικαιώματος, όπως είναι οι άθικτοι, οι ντάλιτ και άλλες ε, μειονότητες. Εάν θέλουμε να εξηγήσουμε τις διακρίσεις λόγω κάστας μόνο με ε, θρησκευτικές ε, ή πολιτισμικές ιδιαιτερότητες ε, προδίδουμε αυτούς που υποφέρουν που είναι και άνθρωποι, άνθρωποι όντω όπως και όλοι μας και δεν αφορά αυτό το φαινόμενο μόνο την Ινδία, είναι ευρέως διαδεδομένο και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα ενταχθεί ε, στη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και το ζήτημα αυτό ε, της ε, κατάργησης των διακρίσεων κατά των αφδικτών. Οι διακρίσεις βάσει εθνικής καταγωγής, ε, φιλετικής καταγωγής, ε, σεξουαλικού προσανατολισμού, ε, κάστας, όλες αυτές τις μορφές διακρίσεις πρέπει να καταργηθούν. Είναι θετικό το βήμα που κάνουμε σήμερα, αλλά πρέπει να κάνουμε και άλλα για αυτά τα 160 και πλέον εκατομμύρια ανθρώπους που πλήττονται από αυτή την κατάσταση για να μπορέσουν μια μέρα να ζήσουν με αξιοπρέπεια απολαμβάνοντας όλα τους τα δικαιώματα. Θα ήθελα λοιπόν για μια ακόμη φορά να απευθύνω έκκληση σε όλα τα θεσμικά όρα της Ένωσης να καταπολεμήσουν τις διακρίσεις με συστηματικό τρόπο και σε όλα τα επίπεδα. Στη στρατηγική ανθρωπινών δικαιωμάτων, στο διάλογο με τις χώρες εταίρους και στο σύμβουλο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Καλώ τους συναδέλφους να υποστηρίξουν το ψήφισμα αυτό, να μην απεμπολίσουμε το δικαίωμα ε, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην αξιοπρέπεια που είναι και στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής ταυτότητας για τη Real Politik, το στόχο μας Real να το θυσιάσουμε. Προέδρο, ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Ξενόμητος των Πρασίνων για 1,5 λεπτό η κυρία Τζιν Λάμπερτ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μιλάω και εγώ ως ε, μέλος του δικτύου υποστήριξη των Ταλίτ στο Ηνωμένο Βασίλειο και βεβαίω υπάρχει δέσμευση για την ε, παρέμβαση στι ε, χώρες της Ανατολική Ασία. Βεβαίως θέλω να υποστηρίξω αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, να αντιμετωπίσουμε τα θέματα των διακρίσεων με βάση την κάστα. Κανένας δεν θα πρέπει να αλλάξει την πίστη του για να γίνεται αποδεκτός από την κοινωνία του. Κανένας δεν θα πρέπει να του αρνούνται το νερό σε μια καταστροφή επειδή δεν είναι στην σωστή κάστα και οποιοδήποτε θα μπορεί να υποφελείται από την εκπαίδευση και να χρησιμοποιεί τα ταλέντα του και κυρίως όταν είμαστε σε μια εβδομάδα που εορτάζουμε και την Διεθνή Μέρα της, της Γυναίκας, του Κοριτσιού, αυτό παίρνει ακόμη περισσότερη σημασία. Έχουμε δει την Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίζει τη, εν μέρη τι διακρίσει αυτέ. Έχουμε δει τα προγράμματα τη να κάνουν τεράστια διαφορά. Αλλά έτσι όπω λένε και οι συνάδελφοι, εκτό αν αυτό, μόνο όταν αυτό θα γίνει τμήμα τη γενικότερη αλλαγή θα μπορέσουμε να, να επηρεάσουμε του ανθρώπου, να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πρέπει όλα αυτά να μην αναφέρονται μόνο στα χαρτιά, να υπάρξει εφαρμογή και να υπάρξει οικονομικό πλαίσιο. Ε, πρέπει να δούμε τα δικά μα κρατημέλη. Το Ηνωμένο Βασίλειο πρόσφατα έβαλε ε, θέματα διάκρισης με βάση την κάστα στην ε, νομοθεσία του περί αντιμετώπισης διακριτικής μεταχείρισης, με, μεταχείρισης και αυτό πρέπει να γίνει σε πρακτικό επίπεδο. Πρέπει λοιπόν να το γνωρίζουμε, να γνωρίζουμε τι γίνεται και στις δικές μας χώρες, καθώς επίσης και στις αξίες που προωθούμε διεθνώς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάμπερτ. Τελευταίος ομιλητής για αυτό το γύρο είναι ο κύριος Μίκαλ Γκούσταυσον ε, της ε, Γκουε, Βόρειας Πράσινης Αριστεράς, ε, πάρα πολύ αποτελεσματικός πρόεδρος Επιτροπής ε, για τα δικαιώματα της γυναίκας και την ισότητα των φίλων. Δύο λεπτά έχετε κύριε Γκούσταυσον. Τι εισαγωγή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Επίτροπε, κυρία Μάλφουμ. Ήταν είναι δύσκολο να λαμβάνει κανεί το λόγο αφού έχουν πει τόσα ωραία λόγια οι συνάδελφοι. Είναι δύσκολο να κάνει κανεί μια παρέμβαση με χαρακτήρα ευγενή. Αλλά θα προσπαθήσω. Ε, είναι απαράδεκτα αυτά που συμβαίνουν και λαμβάνουν χώρα σε πολλέ χώρε. Όταν ε, νερά κορίτσια και γυναίκε είναι τόσο εκτεθειμένε από τον κίνδυνο, μιλάμε για εκατομμύρια γυναίκε στην Ινδία. Με τρίπτυχη διακριτική μεταχείριση, οι οποίε ουσιαστικά δεν έχουν το δικαίωμα ούτε να καταχωρήσουν στο ληξιαρχείο να, τα, παιδιά που έχουν γεννήσει. Μιλάμε λοιπόν για γάμους ε, με τη βία, για θύματα κακομεταχείρισης, για μια, έναν ολόκληρο πληθυσμό, έναν κόσμο που ονομάζονται Dalit και οι οποίοι δεν προστατεύονται με κανένα τρόπο. Νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη τη μπορούν να κάνουν περισσότερα. Όταν ε, έχουν συνομιλίε με τι χώρε αυτέ θα πρέπει να ξεκινήσουν και ένα διάλογο για τα θέματα αυτά. Ξέρω ότι η κυρία Μάλστρομ εδώ έχει μεγάλη αίσθηση ευθύνη και θέλει να κάνει πολλά, αλλά πρέπει να γίνουν ακόμη περισσότερα. Το να συνεργαστούμε με τι διάφορε οργανώσει που υπάρχουν, εκπροσωπώντα την κοινωνία των πολιτών των χωρών αυτών, είναι καθοριστική σημασία. Κυρίω πρέπει να συνεργαστούμε με τι ενώσει που εκπροσωπούν τι γυναίκε, διότι αυτοί έχουν την πείρα και τη γνώση σε αυτό το τομέα. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να βεβαιωθούμε ότι η διακριτική μεταχείριση λόγω της κάστας μπορεί να εξαλειφθεί και θα εξαλειφθεί από κάθε μέρος του κόσμου και από οποιαδήποτε χώρα. Σε ευχαριστώ Μάικλ. Ολοκληρώθηκε ο γύρος των ομιλητών από τις πολιτικέ πολιτικές ομάδες. Περνάμε τώρα ε, στη... στους άλλους συναδέλφους και πρώτος θα λάβει το λόγο δεπτό ο κύριος Γκέι Μίτσελ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Τζολή, η οποία τόνισε το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης λόγω κάστας. Νομίζω ότι είναι σε ε, πολύ, σε πολύ κατάλληλη θέση στο σώμα αυτό για να θέσει ένα τέτοιο θέμα. Όπω είπε και ο κύριο Κάσμαν όμω προηγουμένω, πρέπει να είμαστε πολύ πιο ενεργοί και να έχουμε πολλαπλή δράση κατά των χωρών αυτών που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν έτσι του πολίτε του. Πραγματικά ε, τα μηνύματα τη έκθεση είναι όλα αξιέπαινα. Ιδίω ότι πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θεωρήσει ω μια ξεχωριστή μορφή ε, διακατοική μεταχείριση αυτού του είδου τη διακατοική μεταχείριση που συζητάμε αλλά μαζί με οποιαδήποτε άλλη μορφή διακριτική μεταχείριση που μπορεί να ε, οφείλεται σε θρησκευτικέ πεπιθήσει, ε, φιλετική προέλευση, ε, σεξουαλικέ προτιμήσει και ούτω καθεξή. Οι γυναίκε Ντάλιτ είναι αυτέ που δέχονται τη μεγαλύτερη σεξουαλική βία. Είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένε. Και είναι θύματα εκμετάλλευσης πολλές φορές ε, είναι θύματα σεξουαλικών βασανιστήριων, σεξουαλικής δουλείας, εκμετάλλευσης. Ζούμε πια στον 21ο αιώνα. Είναι κάτι το απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Αυτό το είδος ειδικατική μεταχείριση δεν απαντάτε μόνο στην Ασία. Μίλησα με κάποιον ε, στο Δουβλίνο, ένα νεαρό, τον Ντάμπιν, ο οποίο είναι από την Ασία και ο οποίο μου με παρακάλεσε να θίξουμε το θέμα αυτό. Διότι τέτοιε τάσει υπάρχουν και σε πολλέ περιοχέ τη Ευρώπη. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που η Πρόεδρό μα έλαβε την πρωτοβουλία να το συζητήσουμε αυτό. Ε, Καλώ περιλήφθη το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη, γιατί είναι κάτι που αφορά όλε τι πολιτικέ ομάδε και όλε στηρίζουν την ε, πρόθεση του. Ε, ζητώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, μαζί μα να κάνει ό,τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό και να μην επεκταθούν κι άλλο τέτοιου είδου φαινόμενα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο η κυρία Ζήτα Γκουρμάη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, συνάδελφοι, οι διακρίσει με βάση την κάστα αποτελούν μια δραματική πραγματικότητα για πάνω από 260 εκατομμύρια πολίτε του κόσμου. Ε, και είναι μία από, τα πιο, μία από τις πιο βασικές παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ανάμεσα σε αυτά τα θύματα του κοινωνικού αποκλεισμού, οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι οι πιο ευαίσθητες ομάδες και αντιμετωπίζουν διαφόρων ειδών διακρίσεις και βία, ε, συν την ε, σεξουαλική βία, εκμετάλλευση. Ε, παρά τι ε, νομοθετικέ πράξει που έχουν γίνει και από τι συνδικές και από τι ε, αρχέ του Νεπάλ, η πραγματικότητα είναι πάρα πολύ σκληρή για του Ντάλιτ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα νέο νομικό πλαίσιο, γιατί αυτό που υπάρχει είναι τελείω αβέβαιο. Έχουν υπάρξει κατευθυντήρες γραμμέ από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη, διακρί... για τη διακρίση με βάση την κάστα. Εγώ θα ήθελα να μα πει η Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων πώ μπορεί αποτελεσματικά να πιέσει για την εφαρμογή αυτών. Επίση να υπογραμμίσω ότι αυτό δεν είναι θέμα μόνο των χωρών τη Νοτιοανατολική Ισία οι, γυναίκε οι γυναίκες ε, ουσιαστικά ε, απασχολούνται σε χώρε ε, που τι χρησιμοποιούν για, ε, ως μοντέρνες σύγχρονες σκλάβες. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Ευχαριστώ. Ζήτα, είναι... Σε ευχαριστώ Ζήτα. Για ένα λεπτό τώρα έχει το λόγο ο κύριος Φιλ Μπένιον. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η προφορική ερώτηση είναι καλόδεχούμενη. Δεν είναι η πρώτη φορά που τίθεται το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, οι διακρίσει δηλαδή λόγω κάστα. Και δυστυχώ ούτε θα είναι μάλλον και τελευταία. Καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια ανοιχτή την κατάσταση. Πρέπει ωστόσο να παραδεχθούμε ότι δεν είναι παρικής η που έχει σημειωθεί. Θα πρέπει αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπους που υποφέρουν αυτές τις διακρίσεις καθημερινά να μην τους ξεχνάμε. Στο Μπαγκλαντές για παράδειγμα, οι διακρίσεις αυτές αφορούν ε, και ένα κομμάτι του μουσουλμανικού πληθυσμού, Χιντεβάν, που πολλοί τους ε, ταυτίζουν με τους μουσουλμάνους, αλλά και άλλοι. Επίσης στο Πακιστάν οι Ντάλιτ έχουν περιορισμένη πρόσβαση στη συμμετοχή στα πολιτικά δρόμενα. Και αυτό νομίζω ότι είναι απαράδεκτο. Και πολλοί από αυτούς ε, συνιστούν και θρησκευτική μειονότητα, άρα διπλά ε, υφίστανται διακρίσεις. Δεν ζητώ από την Κομισιόν και την ΕΕΔ να εξαγάγει σήμερα το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ε, με έναν τρόπο ομοιόμορφο προς όλους, αλλά να εξαγάγουμε τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα ως αξίες. Αυτό δεν θα μπορούσε να συνιστά ε, υπεριαλισμό σε καμιά μορφή. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ αγαπητέ συνάδελφοι. Τώρα έχει το λόγο η κυρία Μαρτίν Άντρης για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Καταδικάζω τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων που γίνονται απέναντι σε 260 εκατομμύρια γυναίκε παγκοσμίω που υποφέρουν ε, από τι διακρίσει με βάση την κάστα. Τα συστήματα με κάστες είναι άδικα ε, γιατί μεταχειρίζονται τους ε, ανθρώπους με βάση την ιεραρχία. Θεωρούν ότι κάποιοι είναι ακάθαρτοι, άθικτοι και δεν ανήκουν στην σωστή κάστα και για τους Ντάλιτ ε, πολύ συχνά ε, θεωρούνται οι πιο, ε, τους δίνονται οι πιο επικίνδυνες δουλειές και πολλές φορές τους υποχρεώνουν να εργαστούν, τους αναγκάζουν να ζουν σε ε, εξαιρετική φτώχεια. Θα πρέπει λοιπόν ε, να υπάρξει μια ρήτρα για, την, ε, για τη διακρίση με βάση την κάστα και στις εμπορικές μας σχέσεις με τις χώρες αυτές, αλλά και στις συμφωνίες σύνδεσης. Η Κομισιόν θα πρέπει επίσης να αναλάβει δράση έτσι ώστε να αντιμετωπίσει τις διακρίσεις αυτές και εντός των συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί καμία κοινότητα πουθενά δεν θα πρέπει να εξαιρείται από την νομοθεσία για την ισότητα και από την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ Μαρτίνα. Τώρα για δύο λεπτά έχει το λόγο η κυρία Όμεν Ρόιτεν. Ik stel vast dat er een groot gevoel van overeenstemming is in dit parlement over eh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταλαβαίνω ότι εδώ υπάρχει ευρία συνένεση στο Κοινοβούλιο ω προ την έκθεση που ετοίμασε η κυρία Ζολή. Και πρέπει να πω ότι πραγματικά έχει πολύ σωστά εντοπίσει τι διαστάσει του φαινομένου που μα απασχολεί. Όταν μιλάμε για διακριτική μεταχείριση λόγω τη κάστα, Πρόεδρε, μιλάμε για ολόκληρε ομάδε των πολιτών που λόγω του γεγονότος ότι γεννήθηκαν σε μια συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού πρέπει να είναι στιγματισμένοι για την υπόλοιπη ζωή του και την χάνουν διαφορετική μεταχείριση. Πρόεδρε, αυτό αποτελεί παραβίαση των βασικότερων θεμελιωδών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε ε, ίσα δικαιώματα σε όλους, ανεξιθρησκεία, ε, ελευθερία να πιστεύει κανείς ό,τι θέλει, ελευθερία να εξελιχθεί στη ζωή του. Δεν θέλουμε άνθρωποι να ζουν σε μια κοινωνία με βάση, με διαθρωμένη με βάση τις κάστες ε, και να είναι θύματα φτώχειας. Υπολογίζεται ότι 60 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίω είναι θύματα τέτοιου είδους διακρατικής μεταχειρήσεις. Μιλάμε για ένα φαινόμενο που έχει βαθιές ρίζες σε κάποιες κοινωνίες εκεί όπου απαντάτε ως επιτοπλίστων. Εάν λοιπόν, ακόμη και αν προβλεφθεί νομοθεσία για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, η ατιμορρησία ε, θα παραμείνει γενικευμένη και η διακριτική μεταχείριση λόγω της κάστας θα παραμείνει ως, ως έχει όπως είπε ο κύριος Μίτσελ, εμείς πρέπει να ασκήσουμε όλου του μοχλου πίεση που διαθέτουμε για να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Έχω υποβάλει και εγώ με τη σειρά μου μια σειρά από ερωτήσεις προς την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, διότι πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να μας απασχολήσει αυτό το θέμα σε επίπεδο πρεσβειών, διπλωματικών υπηρεσιών. Όχι μόνο να συζητάμε, να μελετάμε και να συντάσσουμε εκθέσεις για το τι συμβαίνει, αλλά να αναλάβουμε συγκεκριμένη δράση για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου. Στις περισσότερες συμφωνίες μας με τις χώρες αυτές, ε, ξανά και ξανά ανακύπτει το θέμα αυτό. Είναι ένα από τα θεμελιωδέστερα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρέπει λοιπόν κάτι να κάνουμε και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση θα έπρεπε στην ετήσια έκθεσή τη που δημοσιεύεται στον ιστότοπό τη να δημοσιοποιεί τα προγράμματα ε, που εκπονεί και το τι κάνει σε συνεργασία με τις αρχές των χωρών αυτών για να μετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Ευχαριστώ, Ρία. Ο κύριο Σαρνέτ, που υποτίθεται ότι θα είχε μιλήσει εκ μέρου ε, των ε, συντηρητικών μεταρρυθμιστών, δεν ήταν όταν ήταν η σειρά του στην αίθουσα. Ζήτησε όμως να μιλήσει στο τέλος αυτού του γύρου παρεμβάσεων. Δεν τον βλέπω παρόλα αυτά. Άρα θα δώσω το λόγο στους συναντέλγους που ζήτησαν ε, το λόγο στο πλαίσιο της διαδικασίας προσέλκυσης της προσοχής του Προέδρου Κάτς, τι Άι. Σον Κέλλη, καταρχάς, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω είναι σημαντικό να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό σήμερα. Ε, ιδιαίτερος, λόγω των νέων τεχνολογικών μέσων θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε παγκοσμίω να προστατεύουμε τι αξίε και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Άλλωστε, μπορεί η δράση μα να είναι ταχύτερη από ό,τι στο παρελθόν με τι νέε δυνατότητε που έχουμε. Για τι γυναίκε, ε, Ντάλιτ, έχει υποθεί χαρακτηριστικά ότι ισχύει το αποκτήμα ότι κάποιοι γεννιούνται, όλοι γεννούνται ίσοι, αλλά κάποιοι πιο ίσοι από άλλου. Για μένα, η διακριτική μεταχείριση λόγω τη κάστα σημαίνει ότι κάποιες και κάποιοι γεννώνται ε, και αυτή η ανισότητα τους ακολουθεί σε όλη τη ζωή μέχρι το θάνατο. Όπως ε, είπε και ο κύριος Μίτσελ, μιλάμε για δράση που θα μπορούσε να αναπτυχθεί γύρω από, την, ε, από τον τομέα της αναπτυξιακής μας δράσης, της αναπτυξιακής βοήθειας που προσφέρουμε στις χώρες αυτές. Και αυτό πρέπει να έχει γίνει εδώ και χρόνια. Πρέπει λοιπόν να βεβαιωθούμε ότι κάτι θα γίνει στο μέλλον. Ε, Ευχαριστώ Σόμ. Ο Πολ Μέρφυ τώρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν ε, δεν θεωρείς άνθρωπος δεν εφαρμόζεται σε σένα τα ανθρώπινα δικαιώματα, δεν ισχύουν όπως ε, και μια ακτιβίστρια Ντάλιτ από τον Μπαγκλατές ε, γνωστή, αλλά και άλλα 260 εκατομμύρια άνθρωποι που πλήττονται από διακρίσεις λόγω κάστας. Ε, ακούμε τρομακτικές ιστορίες, ανερίθμητοι βιασμοί κοριτσιών που κάνουν ότι δεν βλέπουν οι αστυνομικοί, ιστορία ενός 18χρονου, μιας 18χρονης φοιτήτριας που της επιτέθηκαν με βιτριόλι επειδή αρνήθηκε την προσοχή κάποιων αγοριών κτλ. Βέβαια ε, δεν περιορίζεται στην Ασία το φαινόμενο αυτό και στη Βρετανία έχουμε πονίδιστες ε, προσπάθειες κυβέρνησης να καθυστερήσει, να μπλοκάρει την επέκταση της, ε, του νόμου περί, περί ισότητα, συγγνώμη, θα πρέπει να καταδικαστεί. Βέβαια δεν σταματά ούτε ο αποκλεισμό, ούτε τα βασανιστήρια, ούτε η δουλεία, ούτε η φόνη. Είναι καθημερινή ιστορία αλλά υπάρχουν πολλοί ακτιβιστές ε, που ε, υψώνουν τη φωνή τους και αυτό δείχνει ε, το δρόμο προς τα εμπρός για μια κοινωνία με ισότητα και με κατάργηση όλων αυτών των βαρορτήτων που βιώνουμε σήμερα. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Μέρφη. Δεν μπορώ παρά να υποκύψω στον πειρασμό να σας πω το εξής. Η Επιτροπή Ανάπτυξης έλαβε την απόφαση ε, επέστρεψε από μια διάσκεψη ε, του ΟΗΕ για αναπτυξιακά θέματα. Ήταν και ο Μίτσελ μεταξύ άλλων και άλλοι συνάδελφοι. Δεν θυμάμαι να ε, αναφέρθηκε αυτό το ζήτημα γιατί ίσως δεν θέλαμε να θίξουμε τη μεγαλύτερη δημοκρατία του κόσμου. κάποιο το είπε, κάποιο ομιλητή, αλλά θα πρέπει να αντιδράσουμε. Γιατί απέναντι στην παγκόσμια κοινότητα ε, βλέπουμε ότι επικρατεί η σιγή ενώ όλοι αναγνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό συνιστά τραγωδία και ε, έλλειψη δημοκρατία. Ε, επιτρέψτε μου να κάνω αυτό το σχόλιο. Απλά εμεί οι λίγοι που είμαστε εδώ παρόντε θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μα αυτό το θέμα. Κύριε Επίτροπε, έχετε τώρα το λόγο για να ολοκληρώσετε αυτή τη συζήτηση απαντώντας στις ε, παρεμβάσεις εκ μέρους της Επιτροπής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω το χειροκρότημα για εσά ήταν. Ευχαριστώ τα αξιότιμα μέλη που έφτιαξαν το θέμα αυτό. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα ότι το 2013 το να έχουμε εκατομμύρια ανθρώπων να θεωρούνται ω άθικτοι και να ε, την χάνουν διακριτική μεταχείριση με τον πιο φρικτό τρόπο είναι πραγματικά απαράδεκτο. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν ε, για να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση αλλά και να το αντιμετωπίσουμε. Κάποιοι από εσά είπατε ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδο. Για παράδειγμα, στην Ινδία η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα καθεστώ που προσφέρει κάποιε ποσοστώσει δράση για αυτέ τι κάστε έτσι ώστε να υπάρχει πολιτική εκπροσώπηση καθώ επίση και για πρόσβαση ε, ναι, στην απασχόληση και στην εκπαίδευση και στη δημόσια, ε, στο δημόσιο τομέα. Επίση υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο νέα νομοθεσία για την αντιμετώπιση των διακρίσεων που ξεκίνησε να ισχύει το 2011. Υπάρχει πρόοδο, αλλά υπάρχει βεβαίω και μεγάλο περιθώριο ε, βελτίωσης. Τα υπάρχοντα εργαλεία που έχουμε προσπαθούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό, όπω σα είπα και στο εισαγωγικό μου σχόλιο, για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις πιο ευαίσθητε ομάδε και να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τον διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα με αυτέ τι χώρε. πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε για αλλαγή μέσω των εργαλείων που έχουμε στα χέρια μας. Επίσης, θα δημοσιεύσουμε και την ετήσια έκθεσή μας, όπως ξέρετε, για την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου και του σχεδίου δράσης για τις διακρίσεις, ε, και με, ε, τις διακρίσεις με βάση την κάστα. Και βεβαίως θα το στείλουμε και σε εσάς. Να πω επίσης ότι η, η στάση αυτή ε, προφανώς ε, δεν αλλάζει και αυτή η νοοτροπία δεν αλλάζει εν μία νυχτή. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση ε, και σε αυτές τις χώρες αλλά και εδώ. Και θέλω να συγχαρώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που υπέβαλε αυτή την έκθεση, που έτυχε αυτή η έκθεση υποστήριξη από όλες τις ομάδες ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να εξασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι που όντως τους ξεχνούμε πολλές φορές δεν θα του ξεχνούμε πια και θα, του δοθεί η θέση που του ανήκει στον κόσμο. και έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τι ε, διακρίσει ε, που αντιμετωπίζουν. Η ΥΠΑΤΗ ε, εκπρόσωπο βεβαίω συνεχίζει να, είναι, να έχει δεσμευτεί ότι θα συνεχίσει τι προσπάθειε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, αγαπητή Επίτροπε. Λάβαμε μια πρόταση ψηφίσματο από την Επιτροπή Ανάπτυξη συγκεκριμένα και με αυτή την ανακοίνωση κλείνει η συζήτηση για το θέμα αυτό και η ψηφοφορία θα λάβει χώρα σήμερα από τις 12